Mes chers collègues, il est 10h30, nous allons commencer. Συνάδελφοι, είναι 10 και μισή, πρέπει να ξεκινήσουμε. Cécile, là. Communication de la présidente, les décisions... Ανακοινώσεις της Προέδρου, αποφάσεις Παρακαλώ ησυχία, έχουμε ξεκινήσει. Pardon, Victor, je t'ai nommé sans faire exprès. Allez, des décisions prises par les... Αποφάσεις των συντονιστών στην χθεσινή συνεδρίαση. Έχετε λάβει ε, αντίγραφα των αποφάσεων. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι τις 12.30 θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Επίση, να επίση την προσοχή σα σε ένα κοινό εργαστήρι που θα διοργανωθεί από την Επιτροπή μα και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Χρηματοδότηση των καθαρών και βιώσιμων μεταφορών, ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών». Θα διεξαχθεί στι 4 Δεκεμβρίου. Οι συζητήσει θα επικεντρωθούν στην χρηματοδότηση των υποδομών και των καθαρών και αυτοματοποιημένων μεταφορών. Ο εισηγητής μας είναι ο Βίμ Βαντεκάμπ. Έχετε λάβει με mail την πρόσκληση και το πρόγραμμα. Σας ε, παροτρύνω λοιπόν να είστε παρόντες. Θα περάσουμε τώρα στη ψηφοφορία. Ας ελέγξουμε πρώτα αν υπάρχει απαρτία. Κυρία Μάισνερ. Uh, Ένα διαδικαστικό ερώτημα. Πριν να ψηφίσουμε, έχω να διατυπώσω μια επίσημη καταγγελία. Φαίνεται πω τα ενδιαφέροντά μα μόνο των Ευρωβουλευτών δεν είναι τόσο σημαντικά όσο των άλλων. Ε, νευρίασα, διότι είπαμε για 10 και 30, αλλά για λίγα λεπτά που πρέπει για να προσαρμοστεί εδώ η τεχνολογία να χρειαστεί όλοι να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. πρόσφατα ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη η διαχείριση του χρόνου. Ήμουν Σάντο, ήρθα 10 λεπτά νωρίτερα από την ε, ώρα μου και ε, είχε ήδη συζητήσει το θέμα. Και αυτό για να διευκολυνθούν οι εκπρόσωποι τη Κομισιόν. Κάτι τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, σημειώνω τις παρατηρήσεις σας κυρία Μάισνερ, αλλά ξεκινήσαμε στι 10.30 όχι για να μου κάνετε εμένα το χατήρι, αλλά επειδή αυτό αναφέρεται στην εμείς διάταξη. Και πολλοί προβουλευτέ έφυγαν όταν έληξε η προηγούμενη ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει απαρτία, δεν ε, ε, μπορώ να ξεκινήσω. Δεν μπορείτε να μου προσάψετε λοιπόν ότι ξεκινώ ε, τη συνεδρίαση στην ώρα της. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Εντάξει, υπάρχει απαρτία. Να ξεκινήσουμε ψηφοφορία για την ε, πρόταση κανονισμού ε, για τους κοινού ε, κανόνες εκμετάλλευσης των ενέργειων υπηρεσιών της κυρίας Ταπαρντέλ. Άρχεται η ψηφοφορία. Με ανομαστική κλίση. Le vote est fermé. Pérez. Et le, la confirmation du vote à plus 32. Bravo, Madame Tapardel. Ωραία. Συγχαρητήρια στην κυρία Ταπαρντέλ. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση Βαντεκάμπ για την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές Μεταφορέ. συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 4. Εντάξει λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est Πέρας. Εγκρίνεται. Γιούρι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε την τροπολογία 80. J'ouvre le vote. Je ferme le Ναι, έχετε δίκιο. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Α Ας επαναλάβουμε τη διαδικασία. Attendez, attendez, attendez. Donc si ça marche Δεν ξανακάνουμε μάλλον τη διαδικασία. Εγκρίνεται η τροπολογία. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ίνκο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την Ήτρε 4 Je Πέρας. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Allez, j'ouvre le vote. Je ferme le vote. Et je... Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. J'aimais au vote. Ήτρε 9. Je ferme le vote. Ah, bah voilà, je vous l'avais... Ναι, απορρίπτεται, όπως σας είπα. Amendement 102. 102. Υπέρ. Α, συγγνώμη, 122, λέει ο πρόεδρο. Pourquoi autant de méchanceté? Μα γιατί τέτοια κακία, κύριε Βαντεκάμπ. και Κατά. απόχε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Α ελέγξουμε. Bah, je vérifie. Il a pas de conflit d'intérêt dedans. Απλή επαλήθευση είναι. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Πέρασε απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 129 Je ferme le vote. Πέρας. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 149 Je le vote. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά και 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 165 Je ferme le vote. απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ήτρα 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ήτρα 16 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. και 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι. Ετολογική σκέψη α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 17. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην οτροπική σκέψη σιγματάφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συναστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι επιλογή σκέψη β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε ετελογή σκέψη δ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η λογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο Βαντεκάμπ. Et nous passons directement au rapport Αμέσως ακολουθεί η έκθεση Meyer για τις αντιπροσωπευτικές δράσεις για τη συλλογική προστασία των, ε, των καταναλωτών. Είστε έτοιμες και έτοιμοι. 31 υπέρ. Τροπολογία 31. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται νομίζω εγκρίνεται Ο, έχετε χάσει τον μη των κυρία Ροποζαλών. Όχι. Ωραία. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. όλες μαζί το μπλοκ α υπέρ κατά αποχές εσείς σοσιαλιστές πως ψηφίζετε καλώς εγκρίνεται ή εγκρίνονται είναι τρεις 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπλοκ β υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά α εδώ είναι λίγο περίπλοκο 48 λοιπόν, σε επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται δύο ταυτόσημες τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται μπλοκ C γάμα υπέρ σε γάμα δηλαδή στα ελληνικά κατά αποχές απορρίπτεται δέλτα μπλοκ Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ F ε, σίγμα τάφ δηλαδή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπλοκ G δηλαδή ζ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μα δεν είναι δυνατόν, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρώ αμέσως στην 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπλοκ ήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπλοκ Ι υπέρ κατά Κύριε Κράμερ, δεν είπα ακόμη καν αν έχει ψηφιστεί. Δεν είπα ακόμη, δεν ανακοίνωσα ακόμα το αποτέλεσμα. Θέλετε δηλαδή να την επαληθεύσουμε. Καλά, θέλετε να την ψηφίσετε ηλεκτρονικά πριν να την ψηφίσετε. Καλώς ανοίγω την ψηφοφορία. Block I, η Ι. Πέρας. Εγκρίνεται. Μπράβο κυρία Φώστερ. Προχωρούμε στην 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 απερίφθη κύριε Γκέλλερ. Κύριε Γκάλερ, συγγνώμη. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ακολουθεί το επόμενο μπλοκ J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλώς, επαλήθευση λοιπόν αρχίζει στο, για το μπλοκ J. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, η υπέρ είναι 21 ψήφι. Μπλοκ K, κάπα δηλαδή, υπέρ. Με συγχωρείτε μια στιγμή, λέει πρόεδρος. Α, όχι, αυτό ε, καταπίπτει το μπλοκ K, διότι και το J. Τώρα, δύο ε, τροπολογίες ταυτόσιμες, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνονται. Επαλήθευση κύριε Άντερσεν, για την 77 και 78. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ακόμα και αν κάποιος δεν ψηφίζει, έχει δικαίωμα να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Ή μάλλον ε, ηλεκτρονική. Μάλιστα, εγκρίθηκαν. Καλώς, συνεχίζουμε. Οι δύο που ακολουθούν, 79-80, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ομοίως. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται αυτή. Η ένα καταπίπτει 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 καταπίπτει η 6 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία, το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με ψήφους 21 υπέρ, 14 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Τώρα, ακολουθεί η τελευταία ψηφοφορία. όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Ταπαρδέλ για την ισότητα επιχειρήσεων για επιγραμμικές ε, υπηρεσίες. 5 λοιπόν, ε, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 6 υπέρ. Α, θέλετε παλήθευση για το 97. Καλώς αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 97. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική έξι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας την επαληθεύσουμε την ψηφοφορία αυτή. Μιλώ για την 102. Πέρας. Εγκρίθηκε. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 106. Θέλετε επαλήθευση. Καλώς. 105. Αρχίζει. Πέρας. Απεριφθεί. Ναι, πάντα με πολύ μικρή διαφορά βέβαια. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε αμέσως στην 110 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κύριε Πίπερ, κύριε Βίρκουνεν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, λίγη προσοχή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Α, ναι. 116. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Θέλετε επαλήθευση, έτσι δεν είναι. 115 λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αν θέλετε επαλήθευση. Καλώς. 10. Τροπολογία 10. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρας. Απερίφθη. 119. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές όμως το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψηφοφορία 119 τώρα είναι σαφές τώρα είναι σαφές το αποτέλεσμα εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 165 πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση λοιπόν. 167 αρχίζει. Πέρας. Α, ισοψηφία. Καλώ το είδατε κύριε Βάντεκαμπ. Απερίφθη λοιπόν. Ε, με πολύ, ε, ήταν, είναι προφανέ ότι ήταν, ε, δεν υπήρχε διαφορά. 168 υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα χρειαστεί επαλήθευση. 31. 31. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 32 υπέρ. Αποχές. Δεν είναι σαφές. ...32 κύριε Μαρινέσκου. Δηλαδή γράφεται με 3 και 2 μετά. Καλώς. Επαλήθευση. Πέρας. Πέρας. Τέλος. Απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα χρειαστεί πάλι η παρήθεση. Αρχίζει. Τέλος. Είναι δύσκολη δουλειά μου σήμερα. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι βέβαια. Ας την επαληθεύσουμε. 193. Τέλος. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε παληθεύσουμε 201 201 λέει η πρόεδρος τέλος Εγκρίνεται πράγματι. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν. 43. Πέρας. Εγκρίθηκε. Α, το είχα δει εγώ, λέει η Λοιπόν, 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε επαλήθευση. 203. 203 λοιπόν. Πέρας. Εγκρίθηκε πράγματι. 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε παρήθευση. 44. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση λοιπόν. 46, επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη, κάπως το είχα διαισθανθεί. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207. Επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίθηκε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε επαλήθευση πριν καν να πω το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία για το 47. Πέρας. Εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209-210 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται καλός τσεκ Κύριε δεν βλέπω να μην πιστεύεστε. Εγώ σας λέω ότι εγκρίθηκε. Εγκρίθηκαν. Πέρας. Εγκρίθηκαν. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Εδώ αυτή καταπίπτει. 49 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε το, την 51. Πέρας της ψήφου εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση 53 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος και απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάποιος ζητεί επαλήθευση. Καλώς. Επαληθεύουμε την υπαριθμόν 1. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Επαλήθευση για τις τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Μάλιστα, επαληθεύομαι. Πέρας. Α, εγκρίθηκαν. Είχατε δίκιο κυρία Ταπαρντέλ. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές επαλήθευση λοιπόν 88 πέρας και απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα, στο, μάλλον έκθεση, το σύνολό της με ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας, 34 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Ταπαρδέλ. Η έκθεσή σας εγκρίθηκε. Ας περάσουμε λοιπόν ε, απευθείας ε, τώρα στην ανταλλαγή απόψεων ε, με τον Γενικό Διευθυντή της Eurocontrol, τον κύριο Μπράναν, που θα έρθει εδώ δίπλα μου στο Προεδρείο.

Allez, nous commençons, s'il vous plaît, pour notre dernier point Ας περάσουμε λοιπόν, το τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης για σήμερα. Παρακαλώ, ας σεβαστούμε τον προσκεκλημένο μας. Έχουμε λοιπόν ε, την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Μπρέναν. Όπως ξέρετε είναι νέος Γενικός Διευθυντής της Eurocontrol ανέλαβε φέτος τα καθήκοντά του και θεωρήσαμε χρήσιμο να συνεχίσουμε ε, αυτό το διάλογο με τον Eurocontrol που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα συζητήσουμε την ε, ε, διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας γιατί βλέπουμε ότι αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των μετακινήσεων στην ενέργεια κυκλοφορία σε συνδυασμό και με τις Απαρχαιωμένε υποδομές. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα τη διαχείριση τη ενέργειας κυκλοφορία στην Ευρώπη. Καλώ ήρθατε κύριε Μπρέναν στην Επιτροπή μα. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα, για να μα ε, παρουσιάσετε την κατάσταση. Ξέρω ότι δεν είναι πολλά τα 10 λεπτά, αλλά δώστε, δώστε μας ένα πλαίσιο, σφαδρές γραμμές, τι κάνετε εσείς απέναντι στον αυξανόμενο όγκο εναέριων μετακινήσεων και μεταφορών. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο σκοπός της παρουσίασής μου είναι να ενημερώσω ε, για την τρέχουσα κατάσταση στον έλεγχο και κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Μαρινέσκου, παρόν. Ε, περιμένετε να ακούσετε κάποιε πληροφορίε. Έχει κεντρικό ρόλο η Eurocontrol στη διαχείριση τη ενέργεια κυκλοφορία. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε 11 εκατομμύρια πτήσει. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε το δίκτυο, να συλλέγουμε τις ε, εισφορές Είμαστε ο μόνος οργανισμός που αφορά και την πολιτική και τη στρατηγική αεροπορία και παρέχουμε επίσης στήριξη ε, στα ευρωπαϊκά σώματα. Είμαστε πανευρωπαϊκός οργανισμός, έχουμε 41 μέλη που συμμετέχουν, συν επιπλέον δύο μέλη όπως η Νορβηγία, το Ισραήλ και το Μαρόκο. Όσον αφορά τον έλεγχο ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη, γνωρίζετε όλοι τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, την πρωτοβουλία του 2004, που είχε σκοπό να εξχρονίσει και να ενοποιήσει τον Ευρωπαϊκό ένα αέριο χώρο. Το συνολικό κόστος ανά έτος είναι 10 δισεκατομμύρια και αυτά ε, συλλέγονται όσες φορές από τις αεροπορικές εταιρείε και συλλέγονται από την Eurocontrol. Αν δούμε το σύστημα στην Ευρώπη, Βλέπουμε ότι έχουμε 62 κέντρα ελέγχου αέρης κυκλοφορίας για 11 εκατομμύριο ε, πτήσεις. Αν το δούμε αυτό σε σχέση με τις ΗΠΑ, εκεί υπάρχουν 23 κέντρα ελέγχου αέρης κυκλοφορίας με 15,7 15,7 εκατομμύρια πτήσεις. Λιγότερο παραγωγικό λοιπόν είναι το δικό μας το σύστημα σε σχέση με τις Αμερική παρόλο που υπάρχουν διαφορές, όμως άμα δούμε ε, ότι έχουμε παρόμοιο όγκο πτήσεων, δεν είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί. Αυτό το καλοκαίρι, αν δούμε τις ε, καθυστερήσει που αντιμετωπίσουμε, την περίοδο μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου, δηλαδή πολύ πρόσφατα, είχαμε 9,9 εκατομμύρια πτήσεις στην Ευρώπη, αύξηση κατά 3,7%. Πέμπτος χρόνος της που είχαμε σημαντικές αυξήσεις. Ο στόχος της Επιτροπής για τις ε, καθυστερήσεις οι πτήσεις ε, διαιρούμενες με τις ε, καθυστερήσεις ήταν 0,5 ο στόχος και είμαστε στο 1,86 λεπτά. Αρκετά πιο πάνω από το επιθυμητό όριο. Για να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα, οι καθυστερήσεις είναι διπλάσιες από το 2017 ε, η καθυστέρηση δυναμικότητα 70% υψηλότερο, όσον αφορά τη στελέχωση και τις καθυστερήσεις 187% πιο πάνω. Κυρίως στη Γαλλία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά με πτήσεις από την Ισπανία και την Βαρκελόνη. Κάποια παραδείγματα. Να δούμε τώρα το Σάββατο, 28 Ιουλίου, 5 η ώρα, ε, UTC, αν πετούσατε από το Λούτον και θέλετε να πάτε στην Κέρκυρα, δεν υπήρχε περίπτωση να το πετύχετε, γιατί υπήρχαν τόσα θέματα, κακές καιρικές συνθήκες, ε, απεργίες. Είχαμε μια κατάσταση που ουσιαστικά ήταν αδύνατον το σύστημα να λειτουργήσει. 461 ε, ρυθμίσεις είχαμε σε μεμονωμένες χώρες. Άρα χρειάζεται ένα πιο κεντρικό σύστημα διαχείρισης στην Ευρώπη. Ο στόχος μας για να σα εξηγήσω. Πέρσι είχαμε 1,3 εκατομμύρια καθυστερήσεων, φέτος υπολογίζουμε 19,6 εκατομμύρια. Πάνω από το διπλάσιο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι σαν ένας κουβάς που τον γεμίζουμε και γεμίζει, αλλά άμα πει ένα, μια μικρή, ένα, ένα κέρμα πάνω στο τέλος, θα ξεχυλήσει. Το πρόβλημα πού είναι. έχει πολύ να κάνει με τη Γαλλία. Οι καθυστερήσει είναι 31,8% από τη Γαλλία, 26,7% από τη Γερμανία και τα υπόλοιπα είναι Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά υπάρχουν μεγάλες χώρες όπως η Ιταλία που δεν έχουν καθυστερήσεις όπως και η Πολωνία. Το θέμα εδώ είναι ο πυρήνας της Ευρώπης, ο οποίος είναι κορεσμένος. Αν δούμε τον αντίκτυπο στους επιβάτες, και αν δούμε τις αεροπορικές εταιρείε. η νούμερο ένα εταιρεία, η μεγαλύτερη Ryanair, 30% των πτήσεων καθυστερούνται από τον έλεγχο ανέρης κυκλοφορίες και ο καθυστέρηση είναι 22 λεπτά περίπου. Air France, υψηλό ποσοστό επίσης, 20% με καθυστέρηση, με τουλάχιστον 20 λεπτά καθυστέρηση. Ο μέσος όρος καθυστέρησης είναι 49 λεπτά. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι μία στις τρεις πτήσεις έχει καθυστέρηση και θα είναι τουλάχιστον 49 λεπτά, κάτι που είναι απαράδεκτο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με πέρσι. Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ε, το σύστημα το πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείε. Δηλαδή οι εταιρείε πληρώνουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αν δούμε την Ryanair, την EasyJet, τη Lufthansa, British Airways, Turkish, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που πληρώνουν. Δεν υπάρχει έλλειψη ρευστού. Είναι ο τρόπος διαχείρισης ουσιαστικά που δεν είναι αποτελεσματικός. Συνοψίζοντας την κρίση αυτή των καθυστερήσεων, είχαμε 11 εκατομμύρια πτήσεις, 3,7% επιπλέον, ε, χιλιομετρικός επιβάτης 1,2 δισεκατομμύρια, συν 6% επιπλέον. Οι επιβάτες που α, επηρεάστηκαν ήταν 347 εκατομμύρια, αύξηση κατά 31% και οι καθοδόν καθυστερήσεις από τον έλεγχο ενέργεια κυκλοφορία είναι 19,6 εκατομμύρια, αύξηση κατά 111%. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από πέρσι. Ποιο είναι αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το κόστο των καθυστερήσεων είναι 14,5 δισεκατομμύρια, έχουμε δηλαδή αύξηση κατά 26%. Το κόστος των ακυρώσεων είναι στα 3,4 δισεκατομμύρια, είναι 38%. Έχουμε λοιπόν ένα ε, συνολικό κόστος στην ευρωπαϊκή οικονομία που ανέρχεται στα 17,9 δισεκατομμύρια. Το 1 τρίτο οφείλεται στη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας. Και οι επιβάτες που επηρεάζονται είναι αυξημένη κατά 31%. Υπάρχουν ε, βελτιώσεις προς το περιβαλλοντικό κομμάτι για την περιβαλλοντική απόδοση. Κατά 2,2% υπάρχει βελτίωση κάθε έτος με τη χρήση νέων αεροσκαφών, νέων εξοπλισμό, νέες μηχανές και αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά την κατάσταση. Όμως, αυτό το καλοκαίρι ε, καταφέραμε να ε, διασώσουμε 5 εκατομμύρια λεπτών καθυστερήσεων. Όμως, αυτό αποτελεί περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν δημιουργούμε δυναμικότητα, κάνουμε μεγαλύτερες διαδρομές ουσιαστικά. Όταν πετάμε στα 90.000 πόδια, αυξάνουμε τις καύσεις καυσίμου και αυτό ε, ανεβάζει τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί αν δεν το βελτιώσουμε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε του στόχου μα. Το, μήνυμα που θέλω να δώσω για το 2019 σε εσά είναι ότι η δυναμικότητα θα είναι στα ίδια παιδά, στην καλύτερη περίπτωση. Ίσως από την Γερμανία να έχουμε χαμηλότερα ποσοστά. Η αύξηση 63% καθυστερήσει θα είναι χειρότερε από το 2018 και βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο να ε, έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αναλάβουμε λοιπόν κάποια μέτρα πέρσι για να αντιμετωπίσουμε τις εγκαθυστερήσεις, όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι την βοήθειά σας. Αυτό που χρειάζεται είναι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ο κύριος Μαρινέσκου κάνει λόγο για το SCS3, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές, γιατί αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι μικρές προσαρμογές. Θα πρέπει να εμπλεκούν και υπάρχει υπηρεσιών αεροναυτιλίας, δεν είναι μονάχα δηλαδή μια ομάδα ενδιαφερομένων. Πώς ήταν η πιο α, δύσκολη μέρα φέτος ήταν ε, η 7η Σεπτεμβρίου του 2018. Βλέπετε τη ροή. 7 η ώρα το πρωί και συνεχίζει όλη την ημέρα. Βλέπετε τις ροές από την Τουρκία, από τον κόλπο, αλλά η κεντρική Ευρώπη, ο πυρήνας της Ευρώπης, έχει πάρει φωτιά. Ήταν η πιο δύσκολη μέρη, αλλά δεν είχαμε καθυστερήσεις. Αλλά ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι όλοι ε, όλα τα σημεία ήταν επαρκώς τελεχωμένα, είχαν γυρίσει κοπέ του οι ελεγκτές ενέργεια κυκλοφορίας. Γιατί μπόρεσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε 37.000 πτήσει την 7η Σεπτεμβρίου και όχι στις 11 Ιουλίου που ο κόσμο θέλει να πάει στι κοπέ του. Έχουμε κάνει μια πρόβλεψη για το πώ θα είναι αυτό σε 12 χρόνια. αύξηση 1,9% κάθε χρόνο έχουμε. Έτσι θα είναι η ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Το τρέχον σύστημα δεν θα μπορέσει με τίποτα να στηρίξει 55.000 πτήσει την ημέρα. Θα υπάρξει πρόβλημα στην κινητικότητα, στην οικονομία, σε οτιδήποτε. Είναι κάτι ανέφικτο. Επομένω, αν δεν προβούμε στι θεμελιώδει μεταρρυθμίσει που προτείνει ο κύριο Μαρινέσκου, και που χρειάζεται και την υποστήριξη της Επιτροπής δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Παναλαμβάνω λοιπόν, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας από τη Ρουμανική Προεδρία. Χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, διαχείριση του δικτύου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το υιοθετήσουμε και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον ενέργειο χώρο, να αλλάξουμε το σχέδιο απόδασης, το οποίο θα βασίζεται ουσιαστικά στο αποτέλεσμα. Και δεν θα έχουμε αποτελέσματα αν δεν πληρώσουμε, αν δεν έχουμε καλή απόδοση. Θα, ε, πρέπει να ε, χρηματοδοτούμε μόνο τις ε, τεχνολογίες ΕΖΑΡ και να μην υπάρχει πλέον ε, η παρεμβολή των ε, παρόχων υπηρεσιών αεροστοφυλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση που φυσικά μας προκαλεί λίγο ρίγη. Ρίγο λοιπόν, σε μένα προσωπικά τουλάχιστον, γιατί διαρωτώ κατά πόσο θα μπορέσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση του όγκου των μετακινήσεων με όλε αυτέ τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε εντυπωσιακά τα στοιχεία μας που παρουσιάσατε. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Κύριε Μαρινέσκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρένα. Είναι δεύτερη φορά που είδε αυτή την παρουσίαση. Και η πρώτη φορά θυμάμαι ότι ήταν ε, απίστευτη για μένα. Τώρα είστε ο πρώτο ε, Γενικό Διευθυντή τη Eurocontrol που έρχεται και μα παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο την αλήθεια, την πραγματικότητα όσο έχει και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν όλοι τι γίνεται και να δουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα και οι NSPs κατάλαβαν ότι θα είναι πολύ δύσκολο σε ένα, δύο, τρία χρόνια να συνεχίσουμε έτσι. Μπορεί να το ξέρουν οι συναδελφοί, αλλά πριν από δύο χρόνια πρότεινα μια μελέτη, ένα πιλωτικό έργο για νέα αρχιτεκτονική του εναέριου χώρου. Έχουμε τώρα τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν προχθές. Και θα έχουμε την τελική έγκριση ε, της Επιτροπής Σοφών που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο. Κατά τη γνώμη μου τα συμπεράσματα είναι πραγματικά εξαιρετικά, πολύ καλά, δεν το περίμενα. Με κάποια λοιπόν οργάνωση και με μικρές τροποποιήσεις μπορούμε να αυξήσουμε την ικανότητά μας κατά 30% και στο μέλλον με την τεχνολογία, τη διαλειτουργικότητα κτλ. Μέχρι το 2025 η αύξηση ικανοτήτων μπορεί να υπερβεί το 50% και μάλιστα κατά πολύ. Και αυτό χρειαζόμαστε τώρα, είναι σαφές. Ο Γενικός Διευθυντής σας παρουσίασε την κατάσταση. Ξέρετε ότι υπάρχει η πρόταση που ε, παρεμποδίζεται από το Συμβούλιο. Στο παρελθόν αυτό ήταν εξαιτία του Γιβραλτάρ. Τώρα δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι το ίδιο. Και επειδή υπήρχε αυτό το κόλλημα στο Συμβούλιο, εγώ πρότεινα το πιλωτικό έργο. Όμως, με τους ενιαίους εθέρες χωρίς κανένα κόστος μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 20-30% χωρίς κανένα κόστος, μηδενικό. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πάρουμε τα συμπεράσματα, τα πορίσματα της μελέτης να τα σεγάγουμε στο ΣΕΣ 2 ΣΥΝ και σε 2-3 μήνες να έχουμε νέο κανονισμό. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, θα γίνει το 2024. Αλλά θα είναι πολύ αργά. Γιατί σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση όπω έκανε με δεκάδε άλλε προτάσει. Θα έχουμε τη νέα Επιτροπή το 2020. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μέχρι τότε θα είναι πολύ αργά. Τέλος, κύριε Μπρέναν, μιλήσατε για ένα ε, πρόγραμμα επιδόσεων, performance scheme, ήταν καλό μέχρι τώρα. Μείωσε το φορτίο των δρομολογίων, τώρα όμως ε, πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια. Θα πρέπει τα τέλη αυτά των δρομολογίων να βασίζονται στην ικανότητα. Εκείνοι που δημιουργούν, εκείνοι να πληρώνουν. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Πολύ καλή παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Μας παρουσιάσετε την κατάσταση όσο έχει και ελπίζω μέχρι τις ευρωεκλογέ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρινέσκου. Κυρία Φώστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον Νέιμαν Μπρένεν που ήρθε στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η παρουσίασή σας ε, ήταν ξεκάθαρη και εύληπτη και για τους ευρωβουλευτές. Εμείς βέβαια συναντηθήκαμε πρόσφατα, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Όπως πολύ ορθώς ε, αναφέρατε και όπως είπε και ο κύριος ε, Μαρινέσκου, βρισκόμαστε στο ίδιο μικρό αυτή τη στιγμή για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, γιατί θα συνεχιστούν οι πιέσεις. Συμφωνείτε μαζί μου όμως ότι ενώ η τεχνολογία θα διαρματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού στον έχουμε να κάνουμε με τον κανονισμό ΣΕΣ 2-3 και ό,τι γίνει στο μέλλον, αυτό είναι ένα τμήμα μόνο της λύσης, γιατί θεωρώ ότι ένα από τα βασικά ε, στοιχεία της παρουσίασής σας και με το οποίο συμφωνώ είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί πολύ και η συνεργασία μεταξύ χωρών, όχι μόνο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί φυσικά καλύπτεται μια πολύ ευρύτερη περιφέρεια και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μαρόκο, Ισραήλ, είπατε μερικέ χώρες. Συμφωνείτε λοιπόν ότι και εκείνοι θα πρέπει να βελτιώσουν την διασυνοριακή συνεργασία. Επιπλέον, οι ANSPs, οι πάροχοι ε, έχουν συμβάσεις αλλά δεν ε, πληρούν, δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους ε, με βάση τα συμβολιά της σε ό,τι αφορά τις ε, χρονοθυρίδες και ούτω καθεξής. Μια διευκρίνηση σε αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε σημαντικό πρόβλημα και αυτό είναι εθνικό πρόβλημα ή και εθνικό πρόβλημα. Και τέλος, συμφωνείτε μαζί μου ότι ενώ έχουμε τα διάφορα περιραίοντα τεχνολογικά προβλήματα, υπάρχει και μία πολύ σημαντική πίεση και πάλι αυτό αναπόκειται στα κράτη-μέλη, στις χώρες. Είναι η έλλειψη δυναμικού ικανοτήτων ε, για τα πολύ απλά πράγματα, όπως οι αεροδιάδρομοι ή μάλλον οι διάδρομοι προσγείωσης. Δεν έχουμε αρκετό τσιμέντο. Το έχουμε δει και στο Heathrow, στην Αγγλία, ότι ακόμα και μετά από 20 χρόνια συζητάμε αν θα υπάρξει τρίτος ε, ε, διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης γιατί ακόμα τρέχουμε με υποδομές ε, του 1978. Με ένα μικρό προβληματάκι λοιπόν γίνεται χαμό. Πρέπει λοιπόν και οι εθνικέ κυβερνήσεις να εξετάσουν πολύ πιο σοβαρά το θέμα των υποδομών, το οποίο και αυτό θα βοηθήσει με τη σειρά του εσάς ε, και θα βελτιώσει και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν που επισημάνατε αυτά τα θέματα. Αν μπορείτε να μας μιλήσετε και λίγο για αυτά που σας έθιξα εγώ, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις για να διευκολύνουμε και το δικό σας έργο. Ευχαριστούμε κυρία Φώστερ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μπρέναν για την παρουσίαση. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτα, Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ Ευρωκοντρόλ και ΙΑΣΑ, της οργάνωσης, δηλαδή, του οργανισμού ΕΑΣΑ. Συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας. Δεύτερη ερώτηση. Το γράφημα που το, οργανογράφημα, το οργανόγραμμά σας, συγγνώμη, το οργανόγραμμά σας δείχνει ότι έχετε ε, μέλη από διάφορους κλάδους της, ε, των αέριων μεταφορών. Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα των δράσεων που έχετε αναλάβει για να μειώσετε τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου τον τελευταίο χρόνο. Και τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε αρκετά για τις καθυστερήσεις που ε, υφίστανται οι ε, επιβάτες. Έχετε μετρήσει την απόδοσή σας σε ό,τι φορά τη συμμόρφωση και αντιμετώπιση αξιώσεων των επιβατών εκ καθυστερήσεων και αν ναι, τι είδους απόδοση κατάφερε να έχει η Ευρωκοντρόλ. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ, η κυρία Ματού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Γενικό Διευθυντή για την ε, ε, παρουσίαση, η οποία επιβεβαιώνει ότι το 2018 ήδη έχουμε δυσκολία να αντιμετωπίσουμε το πλήθος των πτήσεων και τις πολλές καθυστερήσεις και ότι θα πρέπει να περιοριστεί η προσφορά. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και έχοντας υπόψη τις μελλοντικέ εξελίξεις και την καθιέρωση του νέου χρόνου αναφοράς υπαριθμών 3. Έχω ερώτηση. Μέτρα που προτείνει η Ευρωκοντρόλ μπορεί να εξηγήσει τι προτείνει ακριβώς για την αντιμετώπιση της αύξησης της κυκλοφορίας που θα οδηγήσει και σε αύξηση των καταμέσων όρων καθυστερήσεων τα επηρεάζουν κυρίως ε, τους χώρους ε, δραστηριοποίησης των Γερμανών και Γάλλων κέντρων, ε, μάλλον εναριών ελεγκτών. Μπορείτε να δημιουργήσετε και νέες εταιρικές συνεργασίες ώστε να εξορροπήσετε τις ελλείψεις χωρητικότητας. Νομίζουμε ότι η υπερβολική επιβολή ε, επιπέδων κόστους ωφέλειας θα οδηγήσει και σε μείωση της απασχόλησης. Έχετε σκεφτεί να συγχωνεύσετε κέντρα εναέριου ελέγχου των χωρών μελών, αλλά μήπως κάτι τέτοιο είναι πρόωρο, δεν θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν τα του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ευχαριστώ κύριε Κλούν. Ευχαριστώ, Έμον, για το ε, μήνυμά σου. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω του χρόνου να μην μας πεις, εγώ σας τα έλεγα. Είναι όμως σαφές και μας έδειξες ποιες είναι οι προκλήσεις και μας είπες και πώς πρέπει εμείς να ασκήσουμε επίσης. Ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό και ελπίζω με την αλλαγή της Επιτροπής και τις εκλογές και όλα αυτά που θα συμβούν ε, θα είναι δύσκολο για εμάς που θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε κάποια πράγματα. Ελπίζω όμως ότι στη Ρουμανική Προεδρία και με την υποστήριξη του κυρίου Μαρινέσκου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο φάκελο αυτό. Είναι σημαντικό να το γνωστοποιήσουμε αυτό και στους ε, πολίτες μας ότι μπορεί να υπάρχουν σύνορα στο έδαφος αλλά στον αέρα υπάρχουν σύνορα. Επίσης για τις ε, προκλήσεις, τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές. Είμαστε σε δύσκολο σημείο καμπής. Κάνουμε μία έκθεση αυτήν την τροπή για τη στρατηγική της Επιτροπής και κάναμε για τη δυναμικότητα και ήταν σαφές και αυτό που είπατε για, το, για την ρύθμιση με βάση τα αποτελέσματα. Και πάλι όμως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μας δώσετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το προς τα που βαδίζουμε και είναι καιρός πλέον να υψώσουμε τη φωνή μας στο θέμα σε αυτό. Ε, έχετε βρει την πόρτα σε αυτή την επιτροπή. Σας ευχαριστώ και πάλι που βρεθήκατε εδώ και για, την, για το έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κλούνα. Ο κύριος Μπρέναν. Κύριε Μπρέναν, μάλλον ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εγώ έχω να σας θέσω μια σειρά ερωτημάτων. Μας μιλήσατε και κρούετε τον κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και ως προς το περιβάλλον, ότι αν δεν υπάρχει συντονισμένη δράση, κατάσταση, ε, θα είναι περισσότερο και από καταστροφική. Μας μιλήσατε και με παρουσιάσατε πολύ ενισχυτικά στοιχεία. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, είπατε, το κόστος των καυσίμων θα είναι 15 έως 25% πάνω. Πολύ είναι αυτό. Και παράλληλα έχουμε και την απίστευτη διεύρυνση ε, των, και αύξηση του όγκου και πτώση των τιμών από την άλλη. Όταν ο κόσμος αγοράζει στήρια με 20 ευρώ, πώς γίνεται να τα ε, συγκεράσουμε όλα αυτά και πώς αυτό συνδέεται και με τη φορολογία. Εγώ Λέω ότι στους ε, κλάδους ε, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ρήπανση θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή της αρχής ο ρηπαίνων πληρώνει. Και γιατί να μην βάλουμε ας πούμε έναν ε, φόρο της κυροζήνης ή μια νέα νομοθετική διάταξη. Δεύτερον, πολύ σωστά τα είπε ο κ. Μαρινέσκου ότι υπάρχει ζήτημα ουσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Εμείς είμαστε υπέρ βέβαια γιατί αν έχουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε και τις ροές. Τα κράτη-μέλη όμως μπλοκάρουν αυτή την προσπάθεια. Τι κάνετε εσείς λοιπόν απέναντι στα κράτη-μέλη. Θα συναντηθείτε μαζί τους, θα τους πείσετε. Γιατί με τα όσα μας παρουσιάσατε, που πραγματικά ε, μα ανοίγουν τα μάτια, αλλά και μας προβληματίζουν πάρα πολύ για την κατάσταση. Μετά ένα σύντομο ερώτημα τι θα γίνει με τον Brexit. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Εσείς, ως Eurocontrol, όταν ε, θα έχετε να κάνετε και με βρετανικές πτήσεις, πώς, τι κάνετε για να ε, διαχειριστείτε αυτό το ενδεχόμενο μη συμφωνίας. Υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης. Ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν το λόγο τώρα για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το αριθμό του κύριου Μαρινέσκου. Για να είμαι δυσκός πρέπει να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος. Καταλαβαίνω ποιος είναι ο ρόλος μας εδώ. ήταν πάντα... Μας στηρίζεται πάντα. 41 τα κρατημέλη που συμμετέχουν στην Eurocontrol. 41. Άρα όλα αυτά γίνονται προ συμφέρον των κρατών μελών, όμω ε, επειδή είναι πανευρωπαϊκό το δίκτυο, περιλαμβάνουμε τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, την ε, Τουρκία. Γιατί όλες αυτές οι χώρες έχουν ε, συμφωνίες στην αεροπορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ιδρυθεί από τις αεροπορικές εταιρείες, όμως ε, η διακυβέρνηση γίνεται από τα κράτη-μέλη. Άρα όλα τα κράτη-μέλη είναι μέλη του οργανισμού μας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όσον αφορά το θέμα της τεχνολογίας που ανέφερε η κυρία Φώστερ, είναι θεμελιώδης οι τεχνολογίας, αλλά δεν είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει πανάκια σε αυτό το θέμα που θα το λύσει το θέμα. πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον σχεδιασμό των δικτύων γιατί η κυκλοφορία ήταν παντού φέτος το καλοκαίρι αλλά πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία. Ένα καλό παράδειγμα η Brussels Airlines. Παρέχουμε στην Brussels Airlines ένα χρονικό διάστημα 90, 90 λεπτών για καθυστερήσεις ή να φύγει τώρα και να πετάει στα 90.000 πόδι, το οποίο είναι καθόλου αποδοτικό. Έχουμε θέματα με το EU261 και τα θέματα του περιβάλλοντος φυσικά. Όσον αφορά ένα περιβαλλοντικό φόρο για τον Ριπένον, ποιος είναι ο Ριπένον, είναι η αεροπορική εταιρεία ή ο ε, πάροχος. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να το αποσαφηνίσουμε. Για μένα λοιπόν το θέμα του σχήματος απόδοσης, του σχεδίου απόδοσης, για να μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε πρέπει να υπάρχει μια α, ισορροπία ανάμεσα στην, στην αποδοτικότητα, την οικονομική πλευρά και τη δυναμικότητα. Αυτό πρέπει να μετράμε. Δεν είναι ότι μπαίνει στο σύστημα, αλλά αυτό που βγαίνει, προκύπτει από το σύστημα. Είναι μια απλή αρχή που έχουμε εφαρμόσει σε κάθε άλλο κλάδο όπως η ηλεκτρική ενέργεια, παραδείγματο χάρη. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω, α, με ρώτησαν τρεις ερωτήσεις. Δράσεις, τι έχουμε κάνει για να βελτιώσουμε το σύστημα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα είναι ευρωπαϊκό σύστημα. Το να υπάρχει ρύθμιση χώρα αναχώρα είναι καλό, αλλά θα πρέπει να τις συνενώσουμε και προθώ την ιδέα της ενίσχυσης της διαχείρισης του δικτύου, του διαχειριστή μάλλον, ο οποίος ορίζεται από το Συμβούλιο των Υπουργών, αλλά θα πρέπει να είναι ένα επιτελείο ουσιαστικά, όπου θα κατευθύνουμε την κυκλοφορία προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθεί. Άρα δεν προτείνω Κάνατε μια ερώτηση για εξυγίανση. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι εφικτό και ότι πολιτικά θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε μια ε, προσέγγιση από πάνω προς τη βάση. Είχαμε την άλλη ε, προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν καταφέραμε πολλά. Οι περιβαλλοντικές πτυχές πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό ανησυχώ, γιατί ο κλάδος έχει μεγαλύτερη επιρροή στο περιβάλλον. Πρώτον, υποστηρίζουμε το πρόγραμμα, το Project Corsair. Δεύτερον, σε κάθε πτήση σχεδιάζουμε την δομή της, τη διαδρομή της πτήσης. Έχουμε και μελέτη αντικ, τύπου για να μειώσουμε το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, να μειώσουμε την χορύπανση. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό όταν υπάρχει πίεση για τη δυναμικότητα. Αν λύσουμε λοιπόν το θέμα της ε, δυναμικότητας, τότε θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα και το περιβαλλοντικό ζήτημα. Το άλλο έχει να κάνει με τα δικαιώματα ε, και τις καταγγελίες στο πλαίσιο του EU 261. Παρέχουμε στήριξη στις εθνικές αρχές, π.χ. στην αρμόδια αρχή του Μαν Βασιλείου, αν θα πρέπει να, φε... να πληρώσει το κόστος η αεροπορική εταιρεία. Δίνουμε τη γνώμη μας για την αιτία της ε, καθυστέρησης, την ταξινομούμε και έχουμε μια στατιστική υπηρεσία που ασχολείται με αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα του Brexit η Eurocontrol έχει ένα προτέρημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αφήσει τη Eurocontrol, γιατί ε, ξεπερνάμε τώρα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ε, αντιθέτως έχουν γίνει και πιο ενεργοί, άρα στο θέμα της ενέργειας κυκλοφορίας θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Το θέμα δυναμικότητας θα λυθεί ε, εν μία ανοιχτή, αν ολοκληρωθούν ε, οι διαδικασίες για το Brexit, μπορεί του χρόνου να μην ε, γυρίσω πάλι εδώ με ένα τέτοιο θέμα Όμω όμως ε, είναι γεγονό ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Ηνωμένο Βασιλείο και σε σχέση με την ΕΑΣΑ έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας, συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Η ΕΑΣΑ είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια. Εμείς υποστηρίζουμε την ΕΑΣΑ. Δεν είμαστε ρυθμιστές ασφάλειας. Τους στηρίζουμε όμως και έχουμε τακτικές συναντήσεις με τον επικεφαλής. Υπάρχουν εθνικές αρχές, υπάρχει η ΆΣΑ, ασφάλειας και μετά υπάρχουμε και εμείς η Eurocontrol. Είναι επομένω λογικό να συνεργαζόμαστε στενά. Από τότε που ανέλαβα το πόστο αυτό, εντατικοποίησα την συνεργασία με την Επιτροπή. Όμω είναι γεγονό ότι αντιμετωπίσουμε μία κρίση του χρόνου το καλοκαίρι θα αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολε καταστάσει. Πρόσφατα σε μια συνεδρίαση όπου μια νέα μητέρα από το Λίτζ με δύο μικρά παιδιά ε, κάνει οικονομίε για να ταξιδέψει στην Ευρώπη και διαπιστώνει ότι έχει πέντε ώρε καθυστέρηση για να πάει στην Μαγιόρκα. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Και Είμαστε πολύ συνυπεύθυνοι και εμεί στη Eurocontrol και η ελληνικέ εταιρείε κυκλοφορία και οι κοινωνικοί εταίροι. Ε, αν δουλεύουν μια ε, εβδομάδα μόνο το καλοκαίρι και παίρνουν τις υπόλοιπες διακοπές τους ε, σε ε, άλλε χρονικέ στιγμέ, τότε θα είναι πιο εύκολο να μην έχουμε θέμα με τη δυναμικότητα. Ελπίζω να απάντησα σε όλε τι ερωτήσει. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας επισκεφτώ. Στο Συμβούλιο Υπουργών στις 3 Σεπτεμβρίου έκανα κάτι παρόμοιο και ζήτησα και τη δική του συμπαράσταση. Είναι καλές προτάσεις από εδώ, αυτές που μας προτείνετε κύριε Μαρινέσκου και είναι καιρός πλέον να, να λάβουμε δράση. Μποκού! Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρέναν. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε που θα μας επιτρέψουν ε, να εμφυσίσουμε πνοή δυναμισμού ε, γιατί είναι και κατεπήγον. Έχει έρθει η ώρα να διαθέσουμε σε αυτούς εργαλεία τα οποία να είναι μεν ισχυρά, να είναι και αποδοτικά, να μπορούν να εφαρμοστούν δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρέναν που προσήλθατε ενώπιον μας και βεβαίως θα σας υποστηρίξουμε και στη συνάντηση του Συμβουλίου στις 3 και σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε να δείχνετε σε ποιο βαθμό είναι ουσιώδης η συνεργασία μας και βεβαίως και κάποια στιγμή να αντιληφθούν και χωρίς μέλη ότι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Συνεχίζει η Πρόεδρος. Λυπούμε τέλος της συνεδριάσεως. Πολύ λυπούμε που είμαι υποχρεωμένη να σα το ανακοινώσω. Ήταν το τελευταίο θέμα αυτό. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου από τι 3 το απόγευμα. Σα ευχαριστώ. Η πρόεδρος ευχαριστεί και του διερμηνείς. Allez, je vous dis à très bientôt. Ωραία. Σα ευχαριστώ. Χαίρετε.